και προγραμμάτων για να μεταφράσουμε ε, στις, στην, ε, νέο κανονισμό Invest EU την επιτυχία που είχαμε με το ΕΦΣΥ. Γι' αυτό χαιρετίζω ε, την θέση του Κοινοβουλίου για το Invest EU που θα μπορέσει να, να παραγάγει το μοντέλο του ΕΦΣΥ. Στο νομικό κείμενο έχουμε καλό ποσοστό. Επίσης η έκθεση προτείνει αλλαγές που θα έχουν περισσότερες επιπτώσεις ε, και θα στηρίξουν και τις αναπτυξιακές τράπεζες. Ο ρόλος μας ως εξωτερικός βραχίωνας επενδυτικός για πάνω από χρόνια έχουμε υποστηρίξει την αναπτυξιακή πολιτική προς άλλες χώρες με ελάχιστο κόστος για τον προϋπολογισμό των ενωσιακών. Ε, προσπαθούμε να αντλήσουμε από τους χρηματοδοτικούς πόρους και για να βοηθήσουμε τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα δέσμευσή μας ε, για προγράμματα εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου έχουμε τομεακή εμπειρογνωμοσύνη. Είμαστε εξωτερικός λοιπόν βραχίωνας, πολύ δραστήριος και θέλουμε να βελτιώσουμε τη ζωή, τις θέσεις εργασίας, τις μικρές και ε, πολύ μικρές επιχειρήσεις και επίσης να βοηθήσουμε στην Αφρική και τις γυναίκες της Αφρικής. Επίσης στη Λατινική Αμερική να υποστηρίξουμε την διπλωματία και επίσης στη γειτονία μας να απαντήσουμε στις προτεραιότητες της ενωσιακές ανάγκες, όπως έγινε για το πακέτο Ουκρανίας. Επίσης, με την πρωτοβουλία ανθεκτικότητας για τα Βαλκάνια, την άμεση γειτονία. Υποστηρίξαμε τα θέματα μετανάστευσης για τις χώρες υποδοχής, τις ε, χώρες προέλευσης και τις ε, χώρες διέλευσης. Υπάρχουν Υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση από διμερείς οργανισμούς για συνεργασία για νέα μέσα χρηματοδοτικά και νέες καινοτομικέ λύσεις. Οι επιχορηγήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο. Η τράπεζα είναι έτοιμη να διευκολύνει και να ε, συντονίσει την πολιτική αυτών που λαμβάνουν τις αποφάσεις με τις αβεβαιότητες που περι, περιβάλλουν ε, την παγκόσμια κατάσταση με τη ρόλο της Κίνας και, το, και τις απειλές ε, για την, για την αντίληψη της πολυμερούς συνεργασίας θα πρέπει να ασχοληθούμε με παγκόσμια θέματα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε χρηματοδοτικό βραχίωνα και χρειαζόμαστε ισχυρή, ε, ισχυρή ΕΤΕΠ. Στην αρχιτεκτονική μετά το 2020 για την χρηματοδότηση εκτός Ευρώπης. Από ό,τι μάθαμε από το ΕΦΣΙ, από το InvestEU, ε, μπορούμε να μεταφέρουμε τα στοιχεία τα οποία μάθαμε ε, στη νέα πραγματικότητα αυτή την ώρα. Ευχαριστώ κυρία Καπέλ που αναφέρατε ε, στο θέμα της διαφάνειας της λογοδοσίας που είναι σημαντικά για τη διαφάνεια ήδη τώρα είμαστε πρώτοι νομίζω σε σχέση με άλλες χρηματοδοτικούς οργανισμούς και προτιθέμεθα να παραμείνουμε τόσο διαφανείς. Ελπίζω ότι τα κράτη-μέλη θα χρησιμοποιήσουν τα ίδια κριτήρια και πρότυπα για τις δανειοδοτικές δραστηριότητες άλλων οργανισμών. Όπως εμείς έχουμε όλο και περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες μας και τις συνέπειες για τους πολίτες. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή για να μετριάσουμε αυτές τις πρακτικές ε, και είμαστε επαγρυπνούμε ούτω ώστε τα χρήματά μας να μην ε, την χάνουν κατά χρήσεως. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ε, θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει όλους μετά τα γεγονότα τα χθεσινά που έδειξαν ποιες θα είναι οι επιπτώσεις εάν αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο αν σταματήσει να είναι μέλος το Ηνωμένο Βασίλειο θα υπάρχουν συνέπειες θεσμικές και οικονομικές. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την υιοθέτηση της γνώμης του Κοινοβουλίου ε, για την, ε, για την ε, τροποποίηση του καταστατικού του ΣΕΤΕΠ και το κεφάλαιο που θα μειωθεί κατά 4 δισεκατομμύρια. Ε, πρόκειται βεβαίως ε, για ένα, κεφάλαιο που πληρώθηκε από τα κράτη-μέλη και αυτό θα μειώσει τη διανοδιωτική μας ικανότητα. Βεβαίως ένα σενάριο τέτοιο δεν ωφελεί κανέναν. Με, ω σημάδι εμπιστοσύνη στην ΕΤΕΠΑ ε, το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει να ενισχύσει και τη βάση την κεφαλαϊκή μετά το Brexit το μερίδιο του Ηνωμένου Βασιλείου θα αντικατασταθεί ε, και θα αυξηθεί η δραστηριότητα. Μερικά κράτη-μέλη προσφέρθηκαν να αυξήσουν την δική τους συνεισφορά. Συνεπώς έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα μπορούμε να έχουμε μια συμφωνία για αντικατάσταση του μεριδίου του Ηνωμένου Βασιλείου για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε την ικανότητα της ΕΤΕΠ ε, για να επιτυγχάνει τους στόχους πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα χάσουμε όλοι αν αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά νομίζω ότι το Κοινοβούλιο, η Κομισιόν προσπαθεί να μειώσει ε, την ζημία στο ελάχιστο. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε εδώ σε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και τώρα από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Επίτροπο κύριο ε, Κατάινεν. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, πρόεδρε της ε, ΕΤΕΠ, Θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Κάπελ, την εισηγήτρια, για την προσπάθεια την οποία έκανε έχει μεγάλη σημασία η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της ΕΤΕΠ. Είναι κομβικός παράγων για την εφαρμογή των πολιτικών μας προτεραιοτήτων. Η τράπεζα είναι απαραίτητος εταίρος για την εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών στο εσωτερικό και εξωτερικό των συνόρων. Η ΕΤΕΠ έχει αποδείξει την δυνατότητά της να επηρεάσει θετικά τους τομείς τους οποίους καλύπτει. Η εφαρμογή και του FC, η πετυχημένη, δείχνει τις νέες δυνατότητες που υπάρχουν ε, και επέτρεψε στην τράπεζα να καλύψει τα κενά τα επενδυτικά τροποποιώντας το επιχειρηματικό της μοντέλο, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η κοινοτομία και οι υποδομές. Η στρατηγική τοποθέτηση της τράπεζας σε κάποιους κεντρικούς τομείς ε, ήταν αντικείμενο των συζητήσεων που έγιναν το 2018 αναμένοντας εν, την αποχώρηση ενός από τους μεγαλύτερους μετόχους του Ηνωμένου Βασιλείου. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για την καταρχήν συμφωνία στην οποία κατέληξαν τα κράτη-μέλη σε σχέση με την επάρκεια την κεφαλαιοχική της τράπεζας. Αυτό δείχνει ακριβώς ότι ε, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική η ΕΤΕΠ και η συμφωνία έτσι θα επιτρέψει την τράπεζα να διατηρήσει το 3α που έχει και το ύψος των επενδυτικών της δυνατοτήτων. Στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό, η ΕΤΕΠ θα παραμείνει βασικός εφαρμοστικός εταίρος. Ε, στα πλαίσια λοιπόν ε, ε, των, της συνεργασίας με τα επιμέρους ταμεία, Έχουμε δημιουργήσει τα προγράμματα στήριξης, τα προγράμματα εφαρμογής, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα ε, και ε, την καταπολέμηση του αποκλεισμού. Νομίζω ότι τα ποσοστά τα οποία θα εγγραφούν στον κανονισμό είναι ικανοποιητικά. Ταυτόχρονα η εμπειρογνωμοσύνη της ε, συγκεκριμένης τράπεζας θα επηρεάσει θετικά και το πρόγραμμα InvestEU. Τώρα για τις εξελίξεις και τη διεθνή συνεργασία για τη γειτονία μετά το 2020 ε, θα μπορέσουν μέσω της ΕΤΕΠ να συνδυάσουν τις επενδυτικές τους δυνατότητες. Η Επιτροπή προτείνει ένα νέο μέσο το οποίο να λειτουργεί στα πλαίσια μιας ανοιχτής αρχιτεκτονικής που χρησιμοποιεί την εμπορνομοσύνη της ΕΤΕΠ των ε, ιδιωτικών πιστοτικών ιδρυμάτων και των αναπτυξιακών εθνικών τραπεζών. Με την τεράστια εμπειρία που έχει η τράπεζα θα παραμείνει ο σημαντικότερος εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εξωτερικές δανειοδοτικές δράσεις στα πλαίσια του επόμενου δημοσιονομικού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει τις συζητήσεις με την ΕΤΕΠ και τα άλλα οικονομικά όργανα έτσι ώστε να καταλήξουμε σε κάποιες ε, θέσεις που θα επιτρέψουν στην ΕΤΕΠ να προβλέπει καλύτερα το τι θα ακολουθήσει μετά το 2020. Δύο επιμέρους θέματα. Πρώτον, κλιματολογικές αλλαγές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υποστηρίζει ε, την φιλόδοξη στάση στον τομέα αυτό της Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Τράπεζας που θέλει να καλύψει τις αποφάσεις της διάσκεψης των Παρισίων. Οι ε, νέες πηγές ενέργειας και η αποδοτικότητα η ενεργειακή είναι βασική στόχη. Τώρα για την συμμόρφωση, ε, ιδιαίτερα στον τομέα της καταπολέμησης της φοροαποφυγής έγιναν σημαντικότατα βήματα τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό απαιτεί νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για τη φοροαποφυγή, ιδιαίτερα στον τομέα των χρηματοδοτικών και επενδυτικών προσπαθειών. Στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με την ΕΤΕΠ και με άλλους ε, εταίρους οικονομικούς ε, βελτιώνοντας και προσαρμόζοντας τις νέες διαδικασίες συμμόρφωσης στο νέο περιβάλλον. Ήδη από το Μάρτιο του 2008 πήραμε μέτρα για την εφαρμογή, την διευκόλυνση μάλλον της εφαρμογής αυτών των νέων απαιτήσεων. Εγώ είμαι ικανοποιημένος από τις συνεργασίες της ΕΤΕΠ με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των τελευταίων γεγονότων στα πλαίσια της συνεργασίας μας. Και γι' αυτό προσβλέπουμε τις προτάσεις ε, της ΕΤΕΠ και για τις μελλοντικές της ε, πολιτικές, ή μάλλον προτάσεις της ΕΤΕΠ και το πόσο θα επηρεάσουν και ο σχεδιασμό των δικών μας πολιτικών στο μέλλον. Ευχαριστώ την εισηγήτρια λοιπόν για μια επακριβέστατη ε, και σε βάθος παρουσίαση της ισχύουσας κατάστασης. Ευχαριστώ. Από πλευράς της ΙΝΤΑ, ε, ο κύριος ε, Πάκετ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θεωρώ ότι η ΕΤΕΠ e e κάνει καλά τη δουλειά της. Και ξέρουμε ότι τεράστια προγράμματα υποδομών, όπω για παράδειγμα ο περιφερειακό τη Ανβέρσα, έχει χρηματοδοτηθεί από την ΕΤΕΠ. Αν μου, επιτρέπετε, αν μου το επιτρέπετε, να επανέλθω στην χρηματοδότηση τη ΕΤΕΠ. Πολύ συχνά είναι μέσω ομολόγων, ε, τα οποία πολλούνται στη διεθνή αγορά ομολόγων. 60 δις πέρυσι, αλλά το 1 τρίτο περίπου είναι σε δολάρια. Το οποίο σημαίνει ότι είμαστε εκτεθειμένοι σε αμερικανικές κυρώσεις δεν μπορεί επιπλέον επι, ε, ε, πλέον να επιλέξει τις επενδύσεις της η ΕΤΕΠ, τις δανειοδοτήσεις της. Και όπως ξέρετε η Αμερική χρησιμοποιεί το δολάριο και για τους δικούς της γεωστρατηγικούς στόχους. Πρέπει λοιπόν να μειώσουμε τη χρηματοδότηση σε δολάρια. Ευχαριστώ. Και τώρα οι ομιλητές από πλευρά των ομάδων. Πρώτα απ' όλα το ΕΛΚ. Ο κύριος Λάγκεν, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κυρία εισηγήτρια. Καταρχάς ευχαριστώ την κυρία Κάπελ. Πολύ καλή δουλειά. Και κύριε Χόιερ, δεν θα πρέπει να σας εκπλήσει το, πόσο, το γεγονός ότι είναι άδεια η αίθουσα, γιατί αυτή τη στιγμή λαμβάνουν χώρα οι συνεδριάσεις όλων των πολιτικών ομάδων για να αποφασίσουν πώς θα ψηφίσουν αύριο. Θυμάμαι ότι και στην ε, συζήτηση με τον πρόεδρο της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ήταν ε, περίπου τόση. Η έκθεση είναι καλή. Η ΕΤΕΠ είναι πολύ σημαντικός θεσμός. Η κυρία Κάπελ και εσείς αναφερθήκατε στα κύρια στοιχεία. Το ΕΛΚ θα ψηφίσει αυτή την έκθεση με την εισηγήτρια κατά τις συζητήσεις επιτύχαμε να ληφθούν υπόψη τα κυριότερα θέματα που μας ενδιέφεραν και βεβαίως η ΕΤΕΠ είναι η μόνη διεθνής ε, τράπεζα που είναι η ιδιοκτησία των κρατών μελών της Ένωσης και που ε, προσαρμόζεται πλήρως με τις προδιαγραφές και τις πολιτικές της Ένωσης. Αυτό είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Χθε είχαμε την απόφαση, ή μάλλον δεν ε, ελήφθη απόφαση για τον Brexit, αλλά ναι, μεν εγώ προσωπικά ελπίζω να εμποδιστεί το Brexit, αλλά είναι καλό που η ΕΤΕΠ έχει κάνει τις αναγκαίες ενέργειες για να ε, μείνει στο επίπεδό του το κεφάλαιό της. Το γεγονό ότι από πλευράς όγκου κεφαλαίων ε, τα οποία δανείζεται είστε μεγαλύτεροι από την Παγκόσμια Τράπεζα, αυτό θα πρέπει να το μάθουν πολύ περισσότεροι συνάδελφοι. Δυστυχώ όμω δεν είναι παρόντε. Ελπίζω τουλάχιστον αύριο να υπάρξει πολύ ευρεία συνένεση. Γιατί στην Επιτροπή ξέρετε ότι οι φιλελεύθεροι και οι σοσιαλιστές, οι κομμουνιστοί και οι πράσινοι, οι φιλελεύθεροι και οι σοσιαλιστές ε, απόσχαν και οι πράσινοι και οι κομμουνιστές ψήφισαν κατά. Και τελικά η έκθεση πέρασε μόνο με τις ψήφους του ΕΛΚ και του ECR. Αυτό δεν είναι όμως η καλύτερη στήριξη που θα μπορούσε να δώσει το Κοινοβούλιο στην ε, ΕΤΕΠ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα για τους σοσιαλιστές ο κύριος Χαουρέγγι Ατόντο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ συμφωνώ με τους επένους ε, για την έκθεση και για την εισηγήτρια. Αλλά να τονίσω τα εξή που θεωρώ πως δεν ε, αναφέρονται επαρκώς στη θέση του Κοινοβουλίου για τη σημασία της ΕΤΕΠ. Γιατί συμφωνώ ότι σίγουρα είναι ένας παγκόσμιος παράγοντας και έχει τεράστια σημασία για την εφαρμογή των πολιτικών και των προτεραιοτήτων και των στόχων της Ένωσης. Οπότε, Είναι σημαντικό να έχουμε αρκετή δράση και στις τρίτες χώρες. Βεβαίως λειτουργούμε σε πολλές τρίτες χώρες, αλλά δεν θα μπορούσαμε να αυξήσουμε τη δανειοδότηση προς τις χώρες αυτές, σε περισσότερες χώρες. Η Ευρώπη λέγεται ότι είναι ήπια δύναμη, δηλαδή ένα μπλοκ που στην εξωτερική της πολιτική είναι αδύναμη, γιατί δεν έχει επαρκή στρατιωτική παρουσία. Όμω η δανειοδοτική μας δραστηριότητα μέσω αυτής τη τόσο σημαντικής τράπεζας, τόσο σημαντική και τόσο μεγάλη, θα πρέπει να παίζει ένα ρόλο στην εξωτερική πολιτική. Και δεύτερον, εφόσον μιλάμε για τρίτες χώρες, η δεύτερη μου σκέψη είναι ακριβώς ότι οι τρίτες χώρες δεν είναι μόνο οι ανατολικοί μας γείτονες. Τρίτες χώρε δεν είναι όλε ανατολικά μας. Υπάρχει υπερβολική, ε, υπερβολικός τονισμός τις γειτονίες και δεν αναφερόμεθα επαρκώς στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική γιατί παίζονται πολλά στην Αφρική και το ξέρουμε. Η ΕΤΕΠ ναι μεν έχει αρχίσει να λειτουργεί στην Αφρική αλλά ιδιαίτερα για την κλιματική αλλαγή πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Και η Λατινική Αμερική είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να κάνουμε περισσότερο στην Κούβα, στην Κολομβία, στην Κεντρική Αμερική. Γιατί η τράπεζα ναι, μεν κάνει πολύ σημαντικά πράγματα σε αυτές τις χώρες, αλλά πρέπει να κάνει περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρος, ECR. Ο κύριος ε, ε, Ζουκ. Ένα λεπτό. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας που αποδεικνύουν ποιος είναι ο ρόλος της τράπεζας αυτής στα πλαίσια της υποστήριξης του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Αναγνωρίζω επίσης τη συνεργασία των τραπεζών με τις εθνικές αρχές για την αποτροπή των φοροαποφυγών, όπως επίσης και των επιθετικών φορολογικών συμφωνιών. Οι δραστηριότητες αυτές είναι συμπληρωματικές με τις δράσεις οι οποίες οφείλουν να αναλαμβάνονται από την κυβέρνηση της Πολωνίας τα τελευταία χρόνια. Σχετικά τώρα με το πρόγραμμα InvestEU, θα πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι η πρώτη τράπεζα η οποία θα πρέπει να είναι καθοριστικά υπεύθυνη για την διαχείριση προγραμμάτων που έχουν ήδη ξεκινήσει να εξελίσσονται. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ επίσης και την κυρία Κάπελ. Και τώρα για την Άλντε, ο κύριος Κόρνιγε. Δύο λεπτά. Κυρία εισηγήτρια, κυρία πρόεδρε, ναι, είναι αδιάψευστο γεγονός ότι η ΕΤΕΠ συμβάλλει στην χρηματοδότηση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός αναφερθήκατε στις διμενείς επιπτώσεις του Brexit. Βεβαίως η έκθεση υπογραμμίζει τον ρόλο των ε, θετικών της ΕΤΕΠ. Θα ήθελα να επισύρω την προσοχή της πάνω ε, σημεία. Βεβαίως δεν πρέπει να συμπεριφέρεστε ως μια ιδιωτική τράπεζα και να καλύπτεται τα κενά χρηματοδότησης. Βεβαίως αναφερθήκαμε σε επενδύσεις σε δολάρια σε σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείε ίσως πέραν των όσων επιθυμούμε, θα πρέπει ίσως να καταπολεμήσετε περισσότερο τη φτώχεια, την κλιματική αλλαγή και να συνεχίσετε την μεταρρύθμιση διακυβέρνησης στις προσπάθειες διαφάνειας όσον σας αφορά και όσον αφορά τους διαμεσολαβητές όσον αφορά την φορολογική απάτη, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα πρέπει να επιγρυπνάτε πάνω στις νέες τεχνικές και λιγμούς που χρησιμοποιούν οι ε, εγκληματίες και θα ήθελα ως αναπληρωτικό μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης να επιτείνετε το ρόλο που έχετε στην ανάπτυξη κυρίως απέναντι στην Αφρική και η προτεραιότητα να χρηματοδοτείτε τα έργα αυτά τα οποία είναι προς όφελος των τοπικών παραγόντων και επιτρέπουν ε, στα κράτη αυτά να έχουν έσοδα φορολογικά για να χρηματοδοτήσουν την οικονομική τους πολιτική. Η έκθεση αυτή είναι ε, υπέρ της Ευρώπης και καλό τους συναδέλφους να την υποστηρίξουν. Ευχαριστώ για τους πρασίνους. Ο κύριος Έχουτ, δύο λεπτά. Καταρχάς, εμείς θα καταψηφίσουμε την έκθεση. Γιατί θα το κάνουμε. Γιατί είχαμε καταθέσει πάρα πολύ κρίσιμες ε, τροπολογίες για τις επιδόσεις της τράπεζας που δεν ελήφθησαν υπόψη στις συμβιβαστικές προτάσεις. Η κριτική που κάναμε δεν περιλαμβάνεται, συνεπώς θα καταψηφίσουμε. Σήμερα όμως θα ήθελα να μιλήσω για το κλίμα και για την προστασία του κλίματος και την συνεκτικότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών. Το Νοέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την μακράν αναμενόμενη στρατηγική της, διευκρινίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι μηδενικός ε, πόλος εκπομπής από το 2050. Κανονικά θα έπρεπε το 2040, γιατί ο τομέας αυτός ε, είναι, θα έλεγα, πολύ σημαντικότατο. Συνεπώς λοιπόν μέχρι το 2040 η υποδομή στον τομέα της ενέργειας θα πρέπει να μην χρησιμοποιεί ορυκτά καύσιμα. Οι επενδύσεις λοιπόν τις οποίες κάνουμε σήμερα θα πρέπει να μας δείχνουν ε, το τι θα κάνουμε και στα 20 χρόνια χωρίς εκπομπές διοξιδίου άνθρακα. Θα πρέπει να απομακρυνθούμε απόλυτα από τα ορυκτά καύσιμα και αυτό δυστυχώς δεν συμβαίνει τώρα υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα από την ε, ΕΤΕΠ που πηγαίνουν στα ορεικτά καύσιμα. Ε, πολλές φορές το επιχείρημα είναι η ασφάλεια στη προμήθεια ενέργειας, αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα επιχείρημα το οποίο είναι αντίθετο με τη μακροπρόθεση στρατηγική μας. Είπατε ότι θα επανεξεταστεί η στρατηγική σας στον τομέα του κλίματος. Αυτό θα πρέπει να το κάνετε κατεπηγόντως. Πώς θα δράσετε πώς θα διασφαλίσετε ότι δεν θα πηγαίνουν επιπλέον επενδύσεις στον τομέα ε, των ορυκτών καυσίμων, γιατί κάθε ευρώ που επενδύεται σήμερα μας απομακρύνει από τον στόχο των μηδενικών εκπομπών το 2050, που υποτίθεται είναι ο στόχος τον οποίο θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι αντιφατικό και θα πρέπει να λυθεί σύντομα. Τώρα για την ΚΟΕ, ο κ. Παπαδημούλης. Δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, και η ευρωομάδα της αριστεράς δεν θα υπερψηφίσει, θα καταψηφίσει την έκθεση. Και ο λόγος είναι ο ίδιος ακριβώς που είπε και ο συνάδελφος Eichhout από τους Πράσινους. Καταθέσαμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, κύριε Λάγκεν, που περίπου μας καταγγείλατε, για να ενισχυθεί η καταπολέμηση της φτώχειας, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής η ενίσχυση της διαφάνειας η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και οι τροπολογίες αυτές που καταθέσαμε δεν έγιναν δεκτές διότι η συγγήτρια προτίμησε που ανήκει στο ΙΕΝΕΦ να φτιάξει μια πλειοψηφία μόνο με το ECR και το EPP. Είναι δικαιωμά Αλλά κύριε Χόγερ, νομίζω ότι και κύριε Κατάινεν αυτή η αίσθηση της αυτάρκειας που ο ένας να συγχαίρει τον άλλον δεν βοηθάει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να γίνει καλύτερη. Όντως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει κάνει καλή δουλειά, αλλά πρέπει να γίνει καλύτερη η δουλειά της. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση υστερεί ακόμη σε επίπεδο επενδύσεων και γιατί η Ευρώπη πρέπει να βοηθήσει και εκτός των συνόρων της για την ανάπτυξη επενδύσεων. Θα σας διαβάσω λίγες λέξεις. Η Ευρωπαϊκή, Κεντρική, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν είχε σαφείς μετρήσιμους στόχους από τους οποίους να προκύπτει η επίτευξη του σκοπού της. Δεν είναι δικά μου λόγια. Τα είπε ο Όσκαρ Χέριξ πριν μόλις ένα χρόνο ως μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κύριε Λάγκεν, κομμουνιστής είναι και αυτός, πράσινος, αριστερός. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τα λέει αυτά. Δεν πρέπει να τα πάρουμε υπόψη μας. Ο κ. Κόμπορν από το e ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Τα αντιαμερικά συναισθήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντικατοπτρίζει αυτή η έκθεση. Είναι μάταιο να φανταζόμαστε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, να ενεργεί σε διάφορες χώρες ε, ή να συγκεντρώνει χρήματα από επενδυτές χωρίς να μετατρέπει ε, συνάλλαγμα από το ένα νόμισμα στο άλλο. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να περιορίσει το κατά πόσο βασίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο σύστημα του δολαρίου. Ε, ποιος είναι ο στόχος όμως, ε, η αντίθεσή μας με την ε, αμερικανική εξωτερική πολιτική και τι θέλουμε να δίνουμε δάνεια στο Ιράν. Το να παραβιάζουμε τα εμπάργκο σίγουρα δεν μας αρκούσε και τώρα θέλουμε και πάλι να παραβιάσουμε τις κυρώσεις των, των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι όμως δεν θα πρέπει να φερόμαστε στον πιο σημαντικό σύμμαχό μας και μετά το Brexit θα είναι καλύτερο μας σύμμαχος το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά του προσφέρουμε ε, μία συμφωνία ε, όχι πολύ καλή για την Βόρεια Ιρλανδία που θα παραμείνει. Διακόπτει η πρόεδρος ε, τον ομιλητή. Πρέπει να προχωρήσουμε. Αν ξεπερνάτε κατά 50% τον χρόνο ομιλία σας, ε, δημιουργείτε προβλήματα για τους άλλους συναδέρφους. Σας ευχαριστώ θερμά. Ο κύριος Jean-Luc Schaffhauser, ένα λεπτό παρακαλώ. Merci, Barbara, pour cet excellent rapport. Ευχαριστώ, Μπαρμπαρά, για αυτή την εξαιρετική έκθεση. Το υπογράμμισαν όλοι. Ωστόσο, εγώ θα απέχω γιατί ε, λόγω του κυρίου Χόιερ σας ε, κατηγορώ ότι δεν είχατε αρκετό θάρρος. Σας κατηγορώ ότι δεν προσαρμόσατε την τράπεζα στην ιδιαίτερη περίπτωση και σας καλώ να λάβετε παράδειγμα από τον Φιλίπ Μάιστατ που είχε έρθει για να φάμε μαζί. Τι πρότεινε, να γίνεται χρηματοδότηση μόνο στις αγορές, όχι να βρούμε χρηματοδότηση στην Κεντρική Τράπεζα μέσω μακροπρόθεσμη χρηματοδότησης προσαρμοσμένη στο κάθε project. Τεράστιες δυνατότητες χρηματοδότησης ανοίγονται έτσι. Επίσης πρότεινε να φτιαχτεί ένα οργανισμός χρηματοδότησης συνδεδεμένος με την ΕΤΕΠ, ώστε ακριβώς να χρηματοδοτούνται τα έργα που δεν είναι της αγοράς σε περιοχές που έχουν φτωχύνει λόγω του ευρώ και έτσι να εναρμονιστεί ο βοράς και ο Νότος γιατί από την εισαγωγή του ευρώ ο Βορράς και ο Νότος της Ευρωζώνης ε, συνεχώς απομακρύνονται. Να ένας τρόπος για να προσαρμοστεί το μέσο στις νέες ευρωπαϊκές προκλήσεις. Σας ευχαριστούμε κύριε Σαφχάουζεν. Ο κύριος Φερνάντες, δύο λεπτά. Sí, buenas noches. Muchas gracias, presidenta señor hoyer el plan juncker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 Ε, ε, κατά τη γνώμη μου, χάσαμε τις δυνατότητες τις αντικυκλικές αυτού του ε, στοιχείου και θα ήθελα να δω πώς θα μπορούσε η ΕΤΕΠ να χρησιμοποιήσει καλύτερα και να το βελτιώσει η ΕΤΕΠ αυτό το αντικυκλικό μέσο που είχε αρχικά στη διάθεσή της. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παπαδημούλη, είχατε πρόβλημα με τη διερμηνία? Όχι, εντάξει, ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Βέτς. Θα ήθελα να πω ότι δεν μπορώ να συμφωνήσω ε, με τους επένους που άκουσα. Η ΕΤΕΠ ε, δίνει ε, γενναιόδωρα δάνεια στην Ουκρανία, για παράδειγμα, σε γεωργικές επιχειρήσεις που ε, κερδίζει έτσι 5,6 δισεκατομμύρια ε, με 1,2 ε, εκατομμύρια δάνειο. Και αντίστοιχα δάνεια στις ντομάτες, στο ηλιέλαιο, στην Ουκρανία. και το MHP, η επιχείρηση MHP έχει λάβει 85 ε, εκατομμύρια ε, και μπορεί να διπλασιάσει την παραγωγή της σε κοτόπουλα χάρη στα δάνεια αυτά ε, και έτσι έχει δημιουργήσει θυγατρικές ε, στην ε, Σλοβακία και με τέτοιου είδους dumping εμείς οι Ευρωπαίοι γεωργοί δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε. Πώς θα πρέπει να επιβιώσει μια οικογενειακή επιχείρηση εφόσον μια ουκρανική επιχείρηση πλημμυρίζει την ευρωπαϊκή αγορά με κοτόπουλα που εκτρέφονται σε κλοβούς. Σας ευχαριστώ κύριε Βάιτς. Ε, σας παρακαλώ όλους να ε, περιορίζεστε στον χρόνο ομιλίας σας. Ένα λεπτό είναι ένα λεπτό. Περνάμε στην ε, διαδικασία Catch the Eye. Τρογεύσκη, παρακαλώ, ένα λεπτό. Θα ήθελα να αναφερθώ στις οικονομικέ δραστηριότητες τη ΕΤΕ, αλλά χωρίς να τι αξιολογήσω γιατί δεν έχω τα σχετικά στοιχεία και δεν ε, γνωρίζω την κατάσταση. Ωστόσο, με ικανοποίηση θα ήθελα να πω ότι η κατάσταση ε, της, είναι, ε, της ΕΤΕ είναι καλή και θα πρέπει να χαιρόμαστε γι' αυτό. Θα ήθελα να κάνω μια έκκληση να δώσετε περισσότερη, μεγαλύτερη ε, πίστη στην, ε, στο κλάδο. Ε, ελπίζω να γίνουν και σχετικές επενδύσεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις, γιατί μέχρι τώρα είναι ισχνός ο όγκος τους. Όσον αφορά την Ουκρανία, είναι σημαντικός μας εταίρος τον οποίο θα έπρεπε να υποστηρίξουμε με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μία ερώτηση εν σχέση με τις ε, προοπτικές, τις μελλοντικές προοπτικές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο. Παρακαλώ. Πρόεδρε, κύριε Χόγερ, θα επαναλάβω αυτά που σας είπα και άλλη φορά. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όσον αφορά την Ελλάδα έχει εξελιχθεί στο βασικό χρηματοδότη ξένων εταιριών προκειμένου κυριολεκτικά να αρπάξουν την ελληνική δημόσια περιουσία. σας θέτω το θέμα της fraport μια εταιρεία που έπρεπε να δώσει 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει 14 περιφερειακά αεροδρόμια. από το 1,2 δις ευρώ τα 968 εκατομμύρια είναι με δάνεια. εσείς ως ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων δώσατε στη fraport 280 εκατομμύρια ευρώ για να γίνουν επενδύσεις στα αεροδρόμια γιατί δεν δίνατε αυτά τα χρήματα προηγουμένως στην εταιρεία που διαχειριζόταν τα αεροδρόμια αυτά στο κράτος να κάνει αυτές τις επενδύσεις. επίσης η τράπεζα αλφα bank έδωσε 280 εκατομμύρια στη fraport. η αλφα bank πήρε από εσάς 100 εκατομμύρια δάνειο. τελικά τι κάνετε χρηματοδοτείτε τις ξένες εταιρείες για να αρπάξουν την ελληνική δημόσια περιουσία ας επενδύσουν αυτές οι εταιρείες όχι με τσάμπα φράγκα όχι τσάμπα επενδυτές. Ευχαριστούμε κύριε Μαριά. Ο κύριος Σανκέλη έχει το λόγο. Δεν χρειάζεται να μιλήσω ολόκληρο λεπτό, θα μιλήσω στην επόμενη έκθεση, αλλά με ενδιαφέρον να άκουσα τρεις ευρωβουλευτές να αναφέρονται ε, στο δολάριο και την εξάρτηση της ΕΤΕΠ από το δολάριο. Νομίζω ότι είναι η τελευταία ευκαιρία ε, και από ε, χρηματοοικονομικής και από πολιτικής πλευράς. Ε, θα πρέπει λοιπόν να πάρουμε θέση στο θέμα αυτό στο εγγύς μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κέλλη. Ο Επίτροπος Κατάινεν έχει το λόγο. Παρακαλώ. Uh, um, Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, ε, πολύ σύντομα τρία στοιχεία τα οποία δεν αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτηση αυτής. Τουλάχιστον δεν αναφέρθηκαν επαρκώ, τα οποία όμως είναι πολύ σημαντικά. Συμβουλευτικέ υπηρεσίες, ε, ε, επιχειρήσεις που σχετίζονται με το κεφάλαιο, που είναι νέο στοιχείο στις ε, ε, εργασίες της τράπεζας και η συνεργασία με εθνικές τράπεζες. Είναι σημαντικά τα θέματα αυτά και όσον αφορά το μέλλον της τράπεζας. Ακούστηκαν κάποιες επικριτικές φωνές, λίγες. Θα ήθελα να θυμίσω σε όλους ότι η ΕΤΕΠ είναι μια τράπεζα που ε, κινείται ανάλογα με τη ζήτηση. Δεν αναγκάζει κάποιον να δανειστεί, αλλά εξυπηρετεί τους πελάτες που έρχονται να ζητήσουν ε, χρηματοοικονομικά μέσα. Η ΕΤΕΠ λοιπόν δεν είναι η πανάκια για όλες τις ασθένειες. Είναι χρηματοδότης που παρέχει και τεχνική βοήθεια. Και όσον αφορά την Ελλάδα, χάρη στην ΕΤΕΠ, μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να λάβουν χρηματοδότηση για ε, τα για τις εργασίες τους. Ε, όλοι γνωρίζετε πόσο έχει δυσκολευτεί η ελληνική οικονομία και για λόγους που όλοι γνωρίζουμε, οι ελληνικές τράπεζες δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αλλά η ΕΤΕΠ μέσω και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και με άλλους τρόπους έχουν βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτές. Η ΕΤΕΠ κάνει πολλά για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Η τράπεζα όμως πρέπει επίσης να γνωρίζει τους κινδύνους που συνδέονται με το κάθε ε, χαρτοφυλάκιο. Έχουμε αυξήσει τη χρηματοδότηση για το μετριασμό τη αλλαγή του κλίματο. Όλα εξαρτώνται όμω από του πελάτε, εάν υπάρχουν βιώσιμα έργα. Η ΕΤΕΠ δεν δημιουργεί πολιτική, είναι ε, το χρηματοοικονομικό σκέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ο κύριος Χόιερ έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μεγάλο το φάσμα των ερωτήσεων και των σχολείων που ακούσαμε και μάλλον δεν θα μπορέσω να απαντήσω σε όλους αμέσως αλλά σας ε, υπόσχομαι ότι το γραφείο μας ε, των Βρυξελών θα απαντήσει σε όλα σας τα ερωτήματα και θα έρθει σε επαφή μαζί σας. Κάποιες φορές δεν είναι μια απάντηση πρακτική, αλλά θα είναι μια πολιτική συζήτηση, όπως για παράδειγμα αυτό το θέμα της πορείας προς τις μηδενικές εκπές άνθρακα. Ε, και, και τη χρήση άνθρακα είναι πολύ σημαντική για την τράπεζα. Όμως η τράπεζα δεν είναι αυτή που χαράζει την πολιτική στην Ένωση. Εμείς συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων και αυτό το κάνουμε μέσω των επενδύσεων άνω των 23 δις τα τελευταία χρόνια ε, και ε, θα πάμε μέχρι τα 100 δισεκατομμύρια από το Παρίσι και μετά για την κλιματική αλλαγή και θα κάνουμε και περισσότερα. Όχι μόνο από την πλευρά των project αλλά και από την πλευρά της χρηματοδότησης, η εφεύρεση, των πράσινων ομολόγων από την ΕΤΕΠ ήταν ένα από τα μεγάλα βήματα ε, της χρηματοπιστωτικής κοινότητας για να αντιμετωπιστούν τα θέματα κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, πρέπει να είμαι σαφής πως έχουμε μεγάλο πρόβλημα διεθνώς όσον αφορά τα στάνταρ και τα κριτήρια. Όταν μιλάμε για το πράσινο ομόλογο, για παράδειγμα, δεν παίρνει κανείς ένα χαρτί το βάφει πράσινο και λέει αυτό είναι πράσινο ομόλογο. Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένη ε, σειρά και ταξινόμηση. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε αυτό και σε διεθνείς ε, διασκέψεις, σε παρουσιάσεις άλλων <laughs> θεσμών έχουμε ακούσει ένα σωρό στοιχεία για τις κλιματικές αλλαγές και για τα σχετικά project. Και θα πρέπει να πάμε λίγο πιο στο βάθος και να δούμε τι ακριβώς είναι το κάθε πράγμα και διαπιστώνουμε πως δεν, δεν έχουμε τα ίδια κριτήρια. Πρέπει να καταλήξουμε σε μια ταξινόμηση που να είναι ε, ε, κατάλληλη για όλα τα ε, διεθνή όργανα. Πρέπει να γίνει αυτή η δουλειά. Έχει γίνει για τα πράσινα ομόλογα σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχει μια διεθνή συμφωνία. Παρόμοια πράγματα χρειάζονται για την βιωσιμότητα, γιατί και εκεί έχουμε την ίδια πρόκληση και πρέπει να αναπτύξουμε τα ίδια τα ίδια στοιχεία και προδιαγραφές γιατί οι αγορές έχουν προχωρήσει πολύ και άρα μπορούμε να έχουμε συγκρισιμότητα. Το επόμενο θέμα έχει να κάνει με την υγεία και την παιδεία και εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό ζητώ την υποστήριξή σας όταν ε, πρόκειται για διεθνείς συμφωνίες για αυτά τα θέματα. Δεύτερη παρατήρηση, μια από τις μεγάλες αλλαγέ τα τελευταία χρόνια είναι ότι με το σχέδιο Juncker ε, ήμασταν σε θέση να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση αυτή τη δεκαετία. Ο αντικυκλικό ρόλο τη ε, τράπεζα που υιοθετήσαμε τότε σε μεγάλο βαθμό έχει κλείσει. Όχι τελείω, αλλά πολλά έχουν γίνει. Έχουμε τώρα την υποχρέωση νομίζω να δούμε λίγο πιο ε, λεπτομερώς και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και του διεθνούς ανταγωνισμού και χάνουμε έδαφος καθημερινά. Εδώ και 15 χρόνια τα κράτη-μέλη της Ένωσης επενδύουν 1,5% του ΑΕΠ λιγότερο ε, ανά στην καινοτομία, έρευνα, ανάπτυξη και παιδεία από ότι οι βασικοί μας ανταγωνιστές στη Βόρεια Αμερική. Κανένας δεν θα πρέπει πιστεύει ότι αυτό δεν σημαίνει απώλεια ανταγωνιστικότητα. και γι' αυτό βλέπω να είναι ιδιαίτερη πρόκληση για την ΕΤΕΠ να συμβάλλει στην καλύτερη χρηματοδότηση της καινοτομία τα επόμενα χρόνια και εννοώ καινοτομία ευρύτερα. Ξεκινά από αυτό, από τους παιδικούς σταθμούς και από τα δημοτικά σχολεία. Να πω και κάτι για την Ευρωπαϊκή Ένωση και, το και την Τράπεζα ως εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δράει και εκτός της Ένωσης και σας ευχαριστώ για τα λόγια σας. Κάποιος μίλησε για ήπια δύναμη. Όμως θα πρέπει να έχουμε και τη σχετική εντολή. Δηλαδή η εντολή εξωτερικού δανεισμού για την ΕΤΕΠ ε, υπόκειται μεγάλη απειλή. Αν περιμένετε να κάνουμε περισσότερα και εγώ ευχαρίστω θα έκανα περισσότερα όχι μόνο στην Αφρική αλλά και στη στρατηγική μα σχέση με τη Λατινική Αμερική και την Ασία για παράδειγμα. Θα μπορούσα να σας δώσω και άλλα παραδείγματα. Ευχαρίστω θα το κάναμε, αλλά αυτό θα σήμαινε ενίσχυση τη εντολή εξωτερικού δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την τράπεζά της. Τέλος, Αφρική. Νομίζω ε, ότι οι Ευρωπαίοι οφείλουν να σκεφτούν πώς έγινε να χρειαστεί η μεταναστευτική κρίση για να καταλάβουμε τις προκλήσεις της Αφρικής. Η Αφρική δεν είναι σημαντική για μας μόνο ως πηγή μετανάστευσης, είναι σημαντική ως στρατηγικός εταίρος για τα επόμενα χρόνια και πρέπει οι αναπτυξιακές μας πολιτικές να μετατραπούν από μια σκέψη ε, δωρητή ε, και ε, ευνοούμενου σε μια σχέση ισοτήμων εταίρων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Χόιερ και Τέλος, έχει το λόγο η συγγήτρια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τις παρεμβάσεις τους, ε, λέγοντας ότι όπως είπε ο κύριος Σόιερ, θα ήταν ε, φταίο για τις ε, τρίτες χώρες να υπάρχει αύξηση του αποθεματικού. Αλλά θα ήθελα επίσης να πω ότι η πρωτοβουλία ανθεκτικότητας για την νότια γειτονία και τα Δυτικά Βαλκάνια έχει αυξηθεί κατά 6 δις μέχρι το 2021. Και ε, προσεχώς θα υπάρξει και μια ειδική στρατηγική για την Δυτική Αφρική. Στους συναδέλφους από την ΚΟΕ θα ήθελα να πω ότι 25% του δανειοδοτικού όγκου της τράπεζας ε, χρησιμοποιήθηκε για διάφορα προγράμματα και ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί. Αλλά για να αλλάξει ριζικά αυτή η λειτουργία θα πρέπει να υπάρξει μια νέα εντολή. Κύριε Χόιερ, είπατε ορθά ότι η ΕΤΕΠ δημιουργεί υπεραξία ε, για τις χώρες μέλη. Ε, τα τελευταία 60 χρόνια πλήρωσε ε, Τρία δισεκατομμύρια για επενδύσεις και πολύ περισσότερο από, από τις φορές των χωρών μελών. Επίσης θα ήθελα να πω στον κύριο Κόμπερν ότι η ΕΤΕΠ, όπως είπε και ο κύριος Λάγκεν, ε, δεν θα χάσει την ισχύ της ε, και μετά το Brexit. Τα υπόλοιπα κράτη θα αντικαταστήσουν το μερίδιο ε, του Ηνωμένου Βασιλείου από το δικό τους αποθεματικό και ορισμένες χώρες θα αυξήσουν τις δικές τους εισφορές θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό αυτό και παρακαλώ για την υποστήριξή σας αύριο. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε εδώ και θα γίνει αύριο, θα εξαχθεί αύριο ψηφοφορία. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη έχουμε την έκθεση του κυρίου Πυρίνσκι. Ετήσια έκθεση 2017 για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία και του Προέδρου, του κυρίου Χόιε, στη συζήτηση αυτή. Κύριε Πυρίνσκη, έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά. Thank Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Χόιε, κύριε Επίτροπε. Όπως είπε και η Πρόεδρος, είναι ε, πολύ θετικό το ότι είστε παρόν κατά την ετήσια συζήτηση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Είχα το προνόμιο από τη θέση αυτή να παρακολουθώ στενά τις εργασίες ε, της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και ως μέλος της Σχετικής Επιτροπής και ως εισηγητής. Και χαίρομαι που σήμερα μπορώ να σας παρουσιάσω μια έκθεση που βασίζεται στη θέση του Κοινοβουλίου προηγουμένων ετών και που βρήκε ευρεία υποστήριξη στην Επιτροπή. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι η έκθεση επισημαίνει ότι οι δραστηριότητες δανειοδότησης ε, της τράπεζας ε, για το 2017 ε, αντιπροσωπεύουν 69,9 δισεκατομμύρια και εξετάζονται οι χρηματικές ροές το 2017 καθώς και το λογιστικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η έκθεση αυτή αναφέρεται σε μια συνεχιζόμενη ανησυχία που έχει να κάνει με τη γεωγραφική κατανομή ε, των δραστηριοτήτων της τράπεζας. Ε, κάτι το οποίο έχουμε αναφέρει επανειλημμένα τα περασμένα χρόνια. Για το έτος αυτό τα δεδομένα ε, δείχνουν ε, το ε, πολύ ανησυχητικό ότι το 2017 το μισό των κρατών μελών έλαβαν το 80% του, των συνολικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ε, τα υπόλοιπα έλαβαν μόλις το 10%. Και το τονίζω αυτό υπό το φως αυτών που ακούσαμε από τον Επίτροπο Κατάινεν και τον Πρόεδρο Χόιερ ε, κατά την προηγούμενη συζήτηση ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι παθητικός παραλήπτης αιτήσεων. Αυτό όμως δεν ανταποκρίνεται στις κανονιστικές υποχρεώσεις της τράπεζας να παίξει ενεργό ρόλο για την ισορροπημένη ανάπτυξη και κοινωνικο-οικονομική και εδαφική συνοχή. Κανείς ε, δεν αμφισβητεί την ανάγκη για καλές επενδύσεις, αλλά ο ρόλος ε, της τράπεζας δεν μπορεί να περιοριστεί ε, στο ρόλο ενός παθητικού παραλήπτη αιτήσεων για δάνεια. Και αυτό τονίζεται στις αιτιολογικές σκέψεις της έκθεσης θα πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να γίνεται αξιολόγηση των αναγκών στους διάφορους τομείς για να κλείσουν επενδυτικά κενά και να εντοπιστεί μια σειρά ευκαιριών για μελλοντικές επενδύσεις. Όσον αφορά τη διακυβέρνηση της τράπεζας που ε, εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, θα ήθελα να τονίσω την ε, προοδευτική ανταπόκριση της ε, τράπεζας ε, που ευθυγραμμίζεται με τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την καλύτερη πρόσβαση στα πρακτικά των συναντήσεων των διαφόρων φορέων της τράπεζας, των διαφόρων σωμάτων της τράπεζας, βελτίωση της διαδικασίας προσφυγής, της τράπεζας και θα ήθελα να επικροτήσω τις αλλαγές που έχουν γίνει. Θα ήθελα όμως να κλείσω επισημένοντας ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικά προβλήματα όσον αφορά την πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων των ε, μελών της ε, Διευθύνουσας Επιτροπής ε, και στο Διευθυντικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο. Και ε, επίσης, όσον αφορά την ε, διαφάνεια κατά την αποκάλυψη ε, των στοιχείων της τράπεζας και την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς. Κυρία Πρόεδρε, έχω υπερβεί τον χρόνο μου κατά 30 ή 40 δευτερόλεπτα. Θα κάνω οικονομία στην τελική μου παρέμβαση. Ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Χόιερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου χαρά να απευθυνθώ στην Ολομέλη για δεύτερη φορά και να συζητήσω ε, το θέμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το τι έκαναν ε, στηρίζοντας την ευρωπαϊκή οικονομία. Ιδιαίτερα θα αναφερθώ στον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων και θα επικεντρωθώ στην εκκριτική έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών για την οποία θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και όσους συνέβαλαν σε αυτή την έκθεση. Τον Ιούλιο 2018 χαιρετήσαμε την εκπλήρωση της υπόσχεσής μας να δώσουμε επιπλέον χρηματοδότηση ε, στο ΕΦΣΙ, στο σχέδιο Juncker ε, είχαμε κινητοποίησει 335 δισεκατομμύρια ευρώ ε, και το ποσό αυτό θα αυξηθεί μέχρι το 2020. Ωστόσο, αυτές ε, οι επιτυχίες ε, δεν θα πρέπει να μας αποκρύπτουν το γεγονός ότι παραμένουν κάποιες προκλήσεις. Συζητήσαμε ορισμένες από αυτές και τις επιπτώσεις του Brexit που είναι προφανής. Η, Επιτροπή της, ε, η έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμών ε, αναφέρεται και σε εσωτερικές προκλήσεις ΕΤΕΠ η ενίσχυση της ε, συνοχής είναι μία από αυτές. Η ΕΤΕΠ παραμένει ε, πρωτοπόρο όσον αφορά τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όσον αφορά τα κριτήρια χρηματοδότησης και την ποιότητα της χρηστής ε, διακυβέρνησης. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, όσον αφορά την πολιτική διαφάνεια τη τράπεζα, η οποία αναθεωρήθηκε το 2015 και θα αναθεωρηθεί το επόμενο έτος και στο πλαίσιο προσπάθειας να απαταχθεί η διαφορά και να αυξηθεί η λογοδοσία. Ε, σε σχέση με το ρόλο μα, ε, παράσχουμε αποτελέσματα όσον αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική, είμαστε μια τράπεζα με υψηλέ ε, προδιαγραφέ και συνεργαζόμαστε με την Όλαφ, τον Ευρωπαϊκό Διαμεσολαβητή και έχουμε συνεχή ανταλλαγή εμπειρία με ΜΚΟ. Λαμβάνουμε τα αιτήματα και τι στάσει του πολύ σοβαρά υπόψη μα και χαιρετήσαμε τα 10 έτη από, την, ε, από τότε που στάθηκε ο μηχανισμός ε, υποβολής καταγγελιών και συνεργασία με τον Ombudsman. Ε, επίσης έχουμε μια νέα πολιτική αποκλεισμού από το 2018 πλήρως ευθυγραμμισμένη με την Κομισιόν. Ε, υιοθετήσαμε έναν αναθερμένο μηχανισμό υποβολής ε, καταγγελιών και οι δημόσιες διαβουλεύσεις είναι σημαντικό κομμάτι εδώ. Ε, είμαστε διατεθειμένοι να αντιμετωπίσουμε μελλοντικές προκλήσεις και να ενισχύσουμε τη χρηστή διακυβέρνηση. Το Διευθυντικό Συμβούλιο συμφώνησε στην εκπόνηση ενός οδικού χάρτη για διάφορες ε, μεταρρυθμίσεις. Τέσσερις διαφορετικές δράσεις θα εφαρμοστούν αυτό το χρόνο. Ε, δεν θέλω να επιστρέψω πάρα πολλές λεπτομέρειες, θα αναφερθώ σε μια ιδιαίτερη πτυχή που αφορά ε, την ετήσια έκθεση αυτού του έτους. Θα ενισχύσουμε την ε, εσωτερική διαχείριση κινδύνων ε, βάσει τριών μοντέλων άμυνας στην εσωτερική δομή της τράπεζας. Και αυτό αφορά και τις τραπεζικές υπηρεσίες. Επίσης, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η τράπεζα πρόκειται να αστικοποιήσει την αναθεώρηση του δεοντολογικού κώδικα, κάτι το οποίο απέτυχε και δική μας ε, Εσωτερική Επιτροπή Ελέγχου. Ε, επίσης θα στεθεί μια ομάδα ε, ε, αξιωματούχων για την αξιολόγηση του κινδύνου. Επίσης την ενίσχυση του Μηχανισμού λήψη Αποφάσεων εκ μέρου του Διευθυντικού Συμβούλου τη ΕΤΕΠ. Επίσης, ε, είμαστε στη συνεχή αξιολόγηση της ε, προσθέμενης ε, αξίας που επιφέρει η τράπεζα. Η, το μοντέλο της προσθετικότητας είναι στο κέντρο της πολιτικής της ΕΤΕΠ. Γιατί εάν δεν μας χρειάζονται, εάν ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να κάνει τη δουλειά μας, στην περίπτωση αυτή περισσεύουμε. Άρα λοιπόν η προσθετικότητα δεν είναι κάτι νέο για μας. Αλλά όσον αφορά το εύση, θέλουμε να δείξουμε ότι αυτό το οποίο κάνουμε είναι πράγματι, πράγματι αυτό το χαρακτήρα διάσταση προσθετικότητας. Ε, θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε κάποιες αστοχίες της αγοράς ή σε συγκεκριμένα προβλήματα. Ε, η αξιοπιστία είναι μια αρχική προϋπόθεση βεβαίως ε, και η ΕΤΕΠ ε, έχει μια απτή συμβολή και υποστήριξη διαδικασιών που έρχονται από άλλες πηγές. Εμείς διευκολύνουμε επιλέξιμα προγράμματα που αφορούν τη δημόσια υγεία, για παράδειγμα, κατά τρόπο που η ίδια η αγορά δεν θα μπορούσε να το πράξει, τουλάχιστον όχι στην ίδια έκταση ή στο ίδιο χρονικό περιθώριο. Η ΕΤΕΠ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την καταμέτρηση της προστατικότητα. και προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τι προσπάθειε μας όσον αφορά την ε, ε, αξιολόγηση των ε, αποτελεσμάτων. Ε, κυρίες και κύριοι, θα συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την ε, μετάβαση προς ένα βιώσιμο κλίμα. Ε, θα υποστηρίξουμε την απασχόληση και θα δράσουμε σαν καταλήκτης για επενδύσεις στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Αναγνωρίζουμε ότι η υποστήριξη της καινοτομίας από τη μία πλευρά και η εμβάθυνση της ολοκλήρωσης από την άλλη ε, δεν ε, βρίσκονται σε αντίφαση γιατί μόνο σε ένα πλήρως ολοκληρωμένο οικονομικό περιβάλλον ε, μπορεί να υποστηριχθεί η κοινοτομία σε όλη την Ευρώπη και μόνο μια καινοτόμα ανταγωνιστική Ευρώπη μπορεί να παράσχει την οικονομική και πολιτική θεμελίωση για βαθύτερη ολοκλήρωση και ένταξη. Υποστήριξη της συνοχής και αύξηση της σύγκλησης παραμένουν πρωταρχές για την τράπεζα. Ε, διαρθρωτικά ε, ε, δάνεια για έργα υποδομής. 26% των δραστηριοτήτων μας ήταν το 2015-2016 και το 2017 το 29% δόθηκε σε περιοχές προτεραιότητας όσον αφορά τη συνοχή. Το 2018 υπερεύει αυτό το στόχο όσον αφορά τις περιοχές ε, ε, συνοχής. Οι κλιματικές δράσεις επίσης